Η επόμενη συνεδρία έληξε η συζήτηση. 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι και από τις 3 μετά το μεσημέρι έως τις 7 μετά το μεσημέρι. Η μερίσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες